dealing with the working machine from here. Okay. This time because the cable was okay. so short. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let us start. I propose to start from test voting. We've got uh, quite... Κύριε και κύριοι, σας προτείνω να συνεχίσουμε. Five proposals, so please... Παρακαλώ, ετοιμαστείτε, να είστε έτοιμοι, γιατί ξεκινούμε. Uh, test voting. Μία δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε. Εκτός αν είναι φύγουμε για διακοπές. Ελπίζω να πείτε όχι. Θα δείξει όμως. Λοιπόν, Everybody has voted. Ψηφίσαμε όλοι. Well, my, my goodness. Everybody has voted. Ψηφίσαμε όλοι. Όχι ακόμα. Πέρας ψηφοφορίας. Ε, καταπληκτική πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε, να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ισχύει ότι έχουμε πολύ σημαντικές ψηφοφορίες. Η συγκεκριμένη είναι η κυρία Σοφία Σακοράφα συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση, στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου. Πρίμα. Ονομαστική ψηφορία, έναρξη ψηφορίας. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σακοράφα. Δεύτερη ψηφοφορία, Όπως και προηγουμένως, προσωρινή συμφωνία βάσει του κανόνα 69 σίγμα ΤΑΦ, όπως και προηγουμένως, ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται επίση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές. Ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, αλλά πετύχαμε πολλά. Συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, επόμενη έκθεση. Κυρία Καμπεθόν Ρουίθ αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 2020 με γνώμονα την ενδιαμέση αξιολόγησή της και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές. Αν πάμε ξανά ε, έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ σηκώστε το χέρι σας. 34. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 46 για τη 46 έτσι πέρας ψηφορίας απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 8. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. 75 πέρας α, απορρίπτεται οι 10 συμβαστικοί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 συμβαστικοί 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1.31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 281 υπέρ. Άμεσο εδώ. Ε, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. 281. Δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1.34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κάποιος ε, ψήφισε δύο φορές ε, ψήφισε μόνο δύο φορές συγχαρητήρια ε, καλό παράδειγμα δίνεται μπράβο και οι δυο σας ευχαριστώ εν πάση περιπτώσει Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15α υπέρ. Κατά. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Να δούμε αν έχουμε την ίδια ψηφορία από την άλλη μεριά όμως. Ε, πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχο για την 68. 68. Άμα δεν σηκώνει το χέρι σα, πέρα ε, για την 68, εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3, την 16 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1,71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 183. 183. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 190 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.58 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2.58 πέρας ψηφορίας απορρίπτεται συμβαστική 26 αποχές εγκρίνεται 74 σε με το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός ελέγχος 274 δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 276 υπέρ. Το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 276 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. 284 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26 β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26 σ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26 δέλτα υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 2.91 υπέρ. Κατά. Να, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2.91. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. 2.92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.93 υπέρ. Κατά. ...2.93 απορρίπτεται. 2.94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.95 υπέρ. Κατά. Αποχές. ηλεκτρονικός έλεγχος. 2.95 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοριάς. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.09 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.07 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 308 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 310 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 312 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 29 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 30 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 3 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εποχές κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 31 υπερ κατα εποχές κατά αποχές εποχές εγκρινεται 3.45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.47 υπέρ. Κατά. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 3.47. 3.47 ψηφίσουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 3.48 υπέρ. Κατά ηλεκτρονικός έλεγχος και την 348. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 349. Κατά. Απορρίπτεται. 350 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά α, εγκρίνεται υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 370 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 372 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 ε, εγκρίνεται η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 9 μάλλον σκέτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική D δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20 για την 20 ψηφίζουμε πέρας ψηφορίας απορρίπτεται Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεν σηκώσετε το χέρι σας. Για την 1 τροπολογία 1. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου. Α, διαδικαστικά, ποιο θέλει το λόγο. Ε, πρόεδρε, από τους πράσινους πιστεύουμε ότι εν γέννη είναι καλή η έκθεση. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδες για το έργο τους. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε λόγω της ε, ατυχούς διατύπωσης όλα αυτά την άμυνα. είμαστε κατά της έρευνας υπέρ της αμήνας. Ε, πρόεδρος, ε, συγγνώμη δεν ήταν διαδικαστικό αυτό, ε, άλλη φορά μόνο για διαδικαστικά. Αυτό ήταν επί της ουσίας. Άλλη φορά δεν θα το επιτρέψω. Ε, είναι ε, σε παράβαση, κατά παράβαση του κανονισμού. Ονομαστική λοιπόν ψηφορία επί του συνόλου του ψηφίσματος. Υπέρ. συγγνώμη, ηλεκτρονική. Συγγνώμη, λέει πρόεδρο. Είναι ηλεκτρονική η ψηφοφορία. Πέρας ψηφορίας. Νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει. Ε, συγχαρητήρια στην κυρία Καπεσόν Ρουίς. Και τώρα. Το αποτέλεσμα. Α, 50 υπέρ. 2 κατά. 5 εποχές. Δεν το είδατε το αποτέλεσμα στην οθόνη μπροστά σα. Ωραία, να το πω τότε. Η κυρία Ματίας ε, έχει κάτι διαδικαστικό. Κυρία Ματίας. Πρόεδρε. Πριν περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία, να ευχαριστήσω όλους τους ασκιώδεις ηγητές. Είχαμε πολλή δουλειά πραγματικά. Ήταν δύσκολη η διαπραγμάτευση, αλλά πιστεύω ότι καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό συμβασμό. Ζήτησα τον λόγο, διότι έχουμε εδώ ένα άρθρο που είναι δική μας αρμοδιότητα και επί του οποίου αντιμετωπίσουμε δυσκολίε, γιατί είχαμε να συγκεράσουμε αντίστάμενε απόψει μεταξύ ΓΚΟΕ, Πρασίνων, ΕΛΚ, Συντηρητικών, TFTD, από την μεριά και σοσιαλιστές από την άλλη. Ήρθαμε εδώ και είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ δύο συμβαστικών τροπολογιών. Αυτά είναι η δημοκρατία, κανένα πρόβλημα σε εκεί. Όμω, στου κοιόδε αποφασίσαμε να μην συμπεριλάβουμε τα παραρτήματα στη ζήτηση, όχι επειδή δεν ήθελα, αλλά επειδή αυτό συμφωνήσαμε από κοινού. Η 6Β, η συμβαστική 6Β των σοσιαλιστών και των φιλελευθέρων ε, συμπεριλάβαν τα παραρτήματα. Εγώ τους είπα ότι δεν ε, θα αντιταχθώ, αλλά θυμίζω για άλλη μια φορά ότι δεν Ψηφίζουμε μεταξύ δύο ισοδυνάμων εναλλακτικών όμω συμβαστικών τροπολογιών. Έχουμε από τη μια μεριά όλε τι πολιτικέ ομάδε, την τροπολογία όλων των πολιτικών ομάδων και η άλλη εναλλακτική τροπολογία ε, των σοσιαλιστών περιλάμβανε τα παραρτήματα, το οποίο, το οποίο όμω δεν περιλάμβανε δική μα τροπολογία, επαναλαμβάνω. Να ξεκαθαρίσω ότι η 6Β περιλαμβάνει, το, ή των σοσιαλιστών περιλαμβάνει τα παρατήματα. Τα, τα λέω όλα αυτά για να υπογραμμίσω για μια φορά ότι δεν είναι ισοδύναμε οι τροπολογίε. μία περιλαμβάνει λοιπόν τα παρατήματα, η άλλη όχι. Παρά τη συμφωνία μα στου Κιώδη. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ για, για το μετριοπαθέ μήνυμα, λέει ο πρόεδρο. Αντιλαμβάνομαι ότι ω ε, εισηγήτρια δεν είστε πολύ ικανοποιημένοι με το χειρισμό του θέματο, αλλά ήταν απόφαση εν τέλει των ε, σκιωδών. Σωστά τα λέτε, η δεύτερη συμβαστική έχει ευρύτερο αντικείμενο σε σύγκριση με την πρώτη, αντίστοιχη συμβαστική. Ε, εδώ δεν έχουμε παράβαση πάντως ε, κανόνα του κανονισμού. Απλώς μας λέτε ότι εσείς ως εισηγήτρια δεν είστε ικανοποιημένοι με την εξέλιξη. Αλλά ότι αυτό ήταν και η απόφαση αν κατάλαβα καλά, από τους σκιώδεις ηγητές. Και η απόφαση αυτή λήφθη εντός προθεσμίας. Ευχαριστώ πάρα για τη δήλωσή σας. Θα τα δούμε αυτά ένα προς ένα κατά τη διάρκεια της ψηφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε ξεκινάμε. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 176 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε την 98. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τα 98. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Συνάδελφε, όταν έχουμε δύο τροπολογίες για το ίδιο ζήτημα, θα ψηφίζουμε τη μία μετά την άλλη. Και αν δεν υπάρχει, αν απορρίπτονται και δύο, θα πρέπει να τις συμφωνούμε, ε, να τις ε, ψηφίσουμε μία προς μία. Οπότε ξεκινούμε. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία της προφορίας εδώ. Οπότε, ας ξεκινήσουμε. Η ε, συμβαστική τροπολογία 6α υπέρ, κατά, άποχες. Ας αρχίσουμε ονομαστική ψηφοφορία, γιατί θα είναι δύσκολο. Λοιπόν, ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 6α. Μάλλον ελέγχουμε για την 6α α. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέραση τη ψηφοφορία απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψήφο για την 6β. Συμβαστική τροπολογία 6β, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία λοιπόν. Πέραση Πέραση Γίνεται δεκτή. 167 λοιπόν. Υπέρ. Στις 167. Κατά αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές γίνεται δεκτή. 151 και 152 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε τη 49 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πέραση της Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές ας την ελέγξουμε ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 55 πέραση της φοφορίας εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 57 ηλεκτρονικά Και την 57 πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε την 60 ηλεκτρονικά. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε την 64. Ηλεκτρονικά λοιπόν για την τροπολογία 64. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 66 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Την 66. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 66. Πέρασε ο Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας. Τροπολογία 4 λοιπόν. Να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 4. Πέρας της 4 εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε την 68 λοιπόν, ηλεκτρονικά. Πέραση της φοφορίας. Εγκρίνεται 69 υπέρ, κατά, αποχές, Ας ελέγξουμε και την 69 ηλεκτρονικά. 69. Πέραση της φοβορίας. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ονομαστική επί του συνόλου. Το Άρχεται ψηφοφορία. ίσως να ψηφίσουμε και μετά σας δώσω το λόγο τη Είναι διαδικαστικό το ζήτημα που θέλετε να θέσετε. Παρακαλώ. Απλώς προφανώς θα καταψηφίσω τη γνωμοδότηση. Δηλαδή αφού υπερψηφίστηκε η τροπολογία 6 και όχι 6α, σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε ε, τη Συμφωνία των Παρισίων, δεν έχουμε δηλαδή μία περίοδο αναφοράς, ξεκινάμε ουσιαστικά από το 0 και δεν ε, αντιμετωπίζουμε επί ίσης όλες, ε, όλες τις χώρες που συμμετείχαν στη διάσκεψη των Παρισιών. Οπότε εμείς θέλουμε να πούμε ότι θα θέλαμε να μείνουμε στο κείμενο της Επιτροπής και να τηρήσουμε αυτήν την ε, Συμφωνία των Παρισίων. Προφανώ ε, ε, εδώ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ψηφίσει κάτι διαφορετικό, κάτι δηλαδή που να αντιώνεται στη Συμφωνία των Παρισίων, αλλά εγώ θα καταψηφίσω αυτό το κείμενο, αυτή την γνωμοδότηση. Πρόεδρο, πέραση τη ψηφοφορία. 44 λοιπόν ψήφοι υπέρ, 13 ψήφοι κατά, μία αποχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία εισηγήτρια. Ευχαριστούμε πολύ τους σκιώδεις εισηγητές και το σύνολο της επιτροπή μας για τις συζητήσεις που έκανε για αυτό το πολύ επίκαιρο θέμα. Περνάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης της κύρια Λόμπες Μπερμέχο σε ό,τι αφορά την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο dumping και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάδελφοι, είναι σημαντικό το θέμα. Έχουμε μια αντίστοιχη κατάσταση εδώ. Δηλαδή, θα έχουμε δύο συμβαστικές τροπολογίες για το ίδιο θέμα. Τη μία μετά την άλλη. Και θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά κάθε φορά. Γιατί το αποτέλεσμα είναι πολύ έτσι κοντά. Η διαφορά είναι μικρή. Θα ψηφίσουμε λοιπόν σημείο προς σημείο. Άμενα κατά των εισαγωγών λοιπόν, έκθεση της κυρία ε, ε Μπεμέχο, 8, συμβαστική, υπέρ. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, λέει ο Πρόεδρος, από την αρχή, κατευθείαν, για τη συμβαστική, 8. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά και πάλι. Γιατί συμβαστική 9. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Γιατί 10. Συμβαστική 10 και πάλι ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Ηλεκτρονικά και πάλι. Πέρας της Εγκρίνεται. Τροπολογίες 58 και 59 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, ας ελέγξουμε λέει πρώτος θα ψηφίσουμε και πάλι ηλεκτρονικά για την 60. Τροπολογία 60, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 12 καταπίπτει. If compromise 10 was not adopted. Not. Oh. Sorry. Yeah. So compromise 10 was not. Η 10 δεν εγκρίθηκε. Οπότε η 12 συμβαστική καταπίπτει. Συμβαστική 13. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και πάλι για τη 13. Συμβαστική τροπολογία 13. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για τη συμβαστική 15. Ηλεκτρονικά. 15. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 75. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 16. Συμβαστική 16. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας για 16. Απορρίπτεται 17 και πάλι ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και πάλι. Για την 6 τροπολογία 6 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Ας ψηφίζουμε και πάλι ηλεκτρονικά, λέει ο για 18. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τροπολογία 18. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 84 υπέρ ξαναρωτάει ο πρόεδρος 84 ένα λεπτό το ελέγχει 84 84 υπέρ κατά αναποχές 86 86 υπέρ κατά απορρίπτεται 87 υπέρ 86 να ελέγξουμε το 86 Ωραία. Για τον 86 λοιπόν ελέγχουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται 87 υπέρ. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 87. 87 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 8. Πέρα τη ψηφοφορία. απορρίπτεται 90 υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται 9 υπέρ. Κατά Αποχέ απορρίπτεται 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά εδώ για τη 12 λέει ο πρόεδρος πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά θα ψηφίσουμε και πάλι ηλεκτρονικά, λέει ο Πρόεδρο, για την 19, συμβαστική 19. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται από ό,τι βλέπω, λέει ο πρόεδρο. Οι σοσιαλιστέ δεν την ψήφισαν. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τα 94, λέει ο πρόεδρο. Είναι ταυτόσιμε. 94 και 95. Τις ψηφίζουμε μαζί. 94 και 95. Ταυτόσιμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ένα λεπτό και πάλι λέει ο πρόεδρο. Τα ξαναλέω λέει ο πρόεδρο. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και θα ψηφίσουμε και για τις 94 95 Πέρα της Αν απορρίπτεται. Σας παρακαλώ, παρακαλώ όμως να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί δεν μπορώ να τα δω λέει ο Πρόεδρος. 96 υπέρ. 96 υπέρ. Ah. Uh, well, could you could you change Αλλάξτε θέση. Και φαίνεται δεν δουλεύει το μηχάνημά σας. Πηγαίνετε προς τα δεξιά σας. Προς τα δεξιά σας, λέει στο κύριο Μπουτικόφερ, ο πρόεδρος. Γιατί δεν δουλεύει το μηχάνημά του. now we go to Ωραία. 96. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 99 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 100 καταπίπτει Πάμε στη 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική 1. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τροπολογία 1. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτή μάλλον, αλλά ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά να δούμε τι γίνεται. Για τη 18 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα τη ε, ψηφοφορία απορρίπτεται 33-22. Η 17 αποσύρθηκε. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και για τη 2. Συμβαστική 2. Πέρα στις ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία 48-12. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε για την συμβαστική τροπολογία 5. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικά και πάλι ψηφίζουμε για τη συμβαστική 6. Άρχεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 6 συμβαστική. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία λέει 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 39 39 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 και 14 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 15 υπέρ, όχι 15 καταπίπτει του λέει ο διπλανός του Πρόεδρου, καταπίπτει 15, συγγνώμη, συγγνώμη, καταπίπτει 15 λέει και ο Πρόεδρος τώρα, γιατί 13 και 14 εγκρίθηκαν. Τελική ψηφορία. Τελική ψηφορία. Πέρα τη ψηφορία. Εγκρίνεται. 30. 30 21 κατά 5 αποχές. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ήταν δύσκολη η ψηφοφορία, αρκετά περίπλοκη όπως είδατε. Έχουμε ένα διαδικαστικό η κυρία εισηγήτρια. Ένα λεπτάκι. Περιμένετε οι υπόλοιποι. Έχουμε την εισηγήτρια ένα διαδικαστικό. Είναι σημαντικό να ακούσουμε. Παρακαλώ καθίστε συναδελφοί. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να πω μόνο ότι προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε μια εναλλακτική που θα προστατεύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και δυστυχώς αυτή η γνωμοδότηση δεν το πετυχαίνει αυτό και θα θέσουμε σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις απασχόλησης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και χρειάστηκε να καταψηφίσω εγώ την ίδια μου την γνωμοδέτηση επειδή ακριβώς δεν προασπιζόμαστε τις θέσεις εργασίας με το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καλωσορίσω τον προσκεκλημένο μας, ο οποίος ευτυχώς έρχεται συχνά στις ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής μας, τον κύριο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Άντρους Άνσιπ αρμόδιο για την ψηφιακή ενέα αγορά έχουμε το επόμενο τμήμα του δομημένου διαλόγου μας και συνεχίζουμε αυτό το διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής και καλέσαμε σχετικά τον κύριο Άνσιπ να μας ενημερώσει για το πρόγραμμα εργασία της Κομισιόν του 2017 που αφορά τις δικέ του αρμοδιότητες. Αλλά και για το 2018 επίσης θα μας μιλήσει. Έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα εργασία της Κομισιόν. Έχουμε εδώ τον κύριο Αντιπρόεδρο, ένα από τους 7 αντιπρόεδρους της Κομισιόν. Θα μιλήσουμε για την πραγματική οικονομία ίσως το ίντερνετ να, είναι, να μην είναι άμεσα πραγματική οικονομία, αλλά την επηρεάζει κατά πολύ. Μα ενδιαφέρει λοιπόν πολύ το πώ ε, προχωράει, το πώ εξελίσσεται η νέα ψηφιακή αγορά. Και αγαπητέ Αντιπρόεδρε, η ψηφιακή ένωση είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, όλες τις επιτροπές μας. Αλλά σήμερα τέλο πάντων θα μιλήσουμε για την ε, νέα ψηφιακή αγορά και το μέλλον της ψηφιακή αγορά και εξελίξεις. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τον Αντιπρόεδρο να μας κάνει την παρουσίασή του. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Το πρώτο είναι πόσα λεπτά έχω. Ο συνήθως 10 λεπτά για την πρώτη σας παρέμβαση. Ε, μετά δεν θα έχετε όμως όριο για τις ε, απαντήσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι κανείς εδώ βεβαίως, αλλά λέει ο Όλοι εδώ θα είναι. Όλοι εδώ θα είναι μέχρι το τέλος. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές της Ήτρε, όπως γνωρίζετε, πριν από δύο χρόνια δρομολογήσαμε τη στρατηγική για την ε, εσωτερική ψηφιακή αγορά. Φέτος, τον Μάιο, προέβημε στην ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής. Υποβάλαμε 35 συνολικά προτάσεις, 21 εξ αυτών είναι νομοθετικού περιεχομένου. Θα ήθελα συνεφώς να πω ότι χάρη στην Επιτροπή σας, την Επιτροπή Ήτρε, η διαδικασία αυτή συνεχίζει. Σημαίνει πρόοδο. Έχουμε καταλήξει σε συμβιβασμούς επιθεμάτων θεμάτων όπως τα 700 MHz. Για παράδειγμα, ένας εξαιρετικά σημαντικός φάκελος, ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Επίσης το 5G στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δίκτυα πέμπτης γενεάς, είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνει πραγματικότητα αν δεν επιλύσουμε το θέμα των 700 MHz. Χαίρομαι όμως, διότι επί αυτού του πολύ σημαντικού θέματος καταφέραμε, επαναλαμβάνω, να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Όσον αφορά τώρα την φορητότητα του ψηφιακού περιεχομένου. Και αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει οι πολίτες μας να έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο όταν ταξιδεύουν στη μια ή την άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρουμε, τουλάχιστον 20% των Ευρωπαίων πολιτών παίρνουν τουλάχιστον 10 μέρες το χρόνο σε κάποια άλλη χώρα. Και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και άλλοι, θέλουν κάθε φορά που ταξιδεύουν να έχουν νόμιμη πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο έχουν αγοράσει. Λόγω διαφορών περιορισμών στο copyright, ώστε δεν μπορούσαν να το κάνουν, όμως χάρη στην παρέμβαση και του Κοινοβουλίου, το οποίο μας υποστήριξε, και μετά από προσπάθηση εννέα μήνων, οι πολίτες μας πλέον έχουν αυτή τη δυνατότητα. Περιαγωγή. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας, γιατί και από αυτού του πολύ σημαντικού θέματος καταφέρουμε να προχωρήσουμε. Το περίμενε ο κόσμος να μπορεί να τηλεφωνά όπως και στη χώρα του. Πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περίμεναν εδώ και 20 χρόνια. Και εδώ, στις περισσότερες περιπτώσεις, το πετύχαμε. Έτσι, η 15η Ιουνίου είναι και το τέλος των τελών περιεγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας ήδη παρέχουν αυτή την ευκολία όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το πεδίο σε όλες τις χώρες. Πρέπει όλοι οι πάροχοι σε όλες τις χώρες να συμμορφωθούν και πρέπει να προσέξουμε να μην σημειωθούν αυξήσεις τιμολογίων με το πρόσχημα της συμπερίληψης της περιαγωγής. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αυξηθούν οι τιμές. Αν θυμάστε, συμφωνήσαμε οι πάροχοι να είναι πολύ προσεκτικοί καθώς ανταλλάσσουν υπηρεσίες. Θέλω λοιπόν να επαγρυπνούμε για κάποιες αυξήσεις, ενδεχόμενες αυξήσεις. Χθε, μάλιστα, συμφωνήσαμε και για την ε, συνθήκη του Μαρακές. Πολύ σημαντικό για τους τυφλούς. Ήταν κρίμα που δεν μπορέσαμε να επικυρώσουμε τη συνθήκη του Μαρακές τα τελευταία τρία χρόνια παρά τον εξελίξη διαθεσμικό διάλογο περί του ποιος δικαιούται να υπογράψει κλπ. Εν τέλει καταλήξαμε, όπως είπα, σε συμφωνία και αυτό θα βοηθήσει πολλούς τυφλούς και ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Κάτι άλλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια καλή είδηση θα έλεγα. Είναι το εξής. επί συγκεκριμένων θεμάτων, πως το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χρειάστηκε να διαπραγματευτούμε το διαδίκτυο των πραγμάτων, η πέμπτη γενεά, κινητή τηλεφωνία πέμπτης γενιάς κλπ. Τα καταφέραμε. Είναι τεχνικά θέματα, αλλά τα καταφέραμε. Χρειάστηκε να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκομένους το θέμα του, της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Ξέρετε, είναι θέματα για τα οποία κάποια κατημέλη λένε μην τα κουμπάτε, είναι εθνική αρμοδιότητα, δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Πάντως πολλοί πρωθυπουργοί και πρόεδροι μας υποστήριξαν σε υπουργικό όμως επίπεδο <laughs> εγγνώμη δίστανται. Έχετε άλλα πέντε λεπτά, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, για το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Χρειάστηκε συνεργασία, επαναλαμβάνω. Χρειάστηκε να θέσουμε και καταληκτικές ημερομηνίες όσον αφορά τις δημοπρασίες για το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Συζήτησαμε τη διάρκεια των αδειών, την κάλυψη αγροτικών περιοχών με δίκτυα πέμπτης γενεάς ή με δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Ε, δεν ήταν ικανοποιητικό το 25, αλλά τέλος πάντων αυτό συμφωνήσαμε εν τέλει, όπως συμφωνήσαμε και θέματα κάλυψης. Τα διασυνδεμένα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Τι θα γίνει με αυτά τα αυτοκίνητα ε, εάν το δίκτυο στην περιοχή δεν είναι πέμπτης γενεάς και επίση συνειδητοποίησαμε και άλλους, τομεί αιστείε, αν θέλετε, τομείς ενδιαφέροντος, την ε, οικονομία των στοιχείων των μεγάλων βάσεων δεδομένων, ελεύθερη διακίνηση δεδομένων, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και εγγυήσει για τις φορολογικές διοικήσεις, για παράδειγμα με τρόπο ώστε να μην στρεβλώνονται τα στοιχεία. Χρειαζόμαστε επίση ηλεκτρονικέ πλατφόρμες που είναι πολύ σημαντικέ για τι συναλλαγέ μεταξύ επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνήθως παραπονούνται διότι δεν έχουν την δυνατότητα να διαπραγματεύονται ισότιμα με τις μεγάλες πλατφόρμες. Πολλές φορές απορρίπτονται από την πλατφόρμα και εκεί ακριβώς εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, αθέμητες επίσης εμπορικές πρακτικές, άλλο ένα θέμα, επιλύση διαφορών. Όλα αυτά είναι θέματα που έχουν σχέση με τις πλατφόρμες. Χρειάζεται επίσης να αποσαφηνίσουμε τα θέματα αναρτήσεων, τα κηρύγματα μίσους, τα οι παραπλανητικές ειδήσει, τα γνωστά fake news και εκεί λοιπόν θέλουμε να βάλουμε μια τάξη στο τοπίο, να ρυθμίσουμε τα κηρύματα μίσους αλλά για όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί συνολικά με τρόπο ενιαίο προστατεύοντας φυσικά την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του λόγου όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να μπορούμε να επεμβαίνουμε σε περιπτώσεις καταγγελιών και να αναλαμβάνουμε δράση. Τι γίνεται όταν κάποιος ανεβάσει περιεχομένο σε μια πλατφόρμα και ε, κάποιος άλλος το αφαιρέσει. Πού είναι τα δικαιώματά μου, πώς προστατεύομαι εγώ πώς προστατεύω τα ένομα συμφέροντά μου, αποκαθιστώντας δηλαδή το περιεχόμενο αυτό στην πλατφόρμα. Και βεβαίω η προστασία στον κυβερνοχώρο χρειάζεται και εδώ να προστατεύσουμε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ενδιαμέσης αναθεώρησης στο πλαίσιο της αναθεώρησης της στρατηγικής αποφασίσαμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ούτω ή άλλω είχαμε ξεκινήσει και το 2013, αλλά από τότε ε, αντιμετωπίσαμε φαινόμενα, ε, ιούς, ε, κακόβουλο, λογισμικό κλπ. που δεν τα είχαμε εκείνη την εποχή. Τα στα botnet, τα οποία μολύνουν σε δεμένες συσκευέ το διαδίκτυο των πραγμάτων, το Internet of Things όπως λέμε. Έχουμε επίση ε, το denial of service, την καταστροφή υπηρεσιών κλπ. Την καταστροφή της πρόσβασης. Αυτές είναι οι προκλήσεις στον κυβερνοχώρο. Πολύ σημαντικές, πολύ σημαντικά προβλήματα, πολύ σημαντικές προκλήσεις. Και εδώ λοιπόν Πρέπει να ενισχύσουμε τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες, να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να την ενισχύσουμε, να την θωρακίσουμε εναντί επιθέσεων όπως οι πρόσφατες. Αυτές στρέφονται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν το σύνολο της. Αυτή τη στιγμή 30 άτομα απασχολούνται 24 ώρες το 24ωρο στην προσπάθειά τους να εξεύρουν ε, λύσεις προστασίας. Στο πλαίσιο λοιπόν του πολίτους δημοσιονομικού προγράμματος πρέπει να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε πόρους και για την κυβερνοασφάλεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος μόνο χρήματα των φορολογουμένων θα αξιοποιηθούν και σε πολιτιακό και σε ομοσπονδιακό επίπεδο για την προστασία 19 δισεκατομμύρια συνολικά. Παρακαλώ. Εμείς θα επενδύσουμε 450 εκατομμύρια από τα χρήματα των φορολογουμένων στο πλαίσιο ΣΔΙΤ για την προστασία του διαδικτύου. Και θα προσθέσουμε σε αυτό 1,8 δισεκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια. Βέβαια οι Αμερικανοί δεν πάρουν ήδη πολύ περισσότερα, αλλά ε, σίγουρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ε, για την κυβερνοασφάλεια, όπω είπα, την ασφάλεια στον χώρο του διαδικτύου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Λεπρόεδρο. Ήσασταν πολύ σύντομο. 13 λεπτά σχεδόν. Μια χαρά είμαστε, λέει ο πρόεδρος, για αρχή τουλάχιστον. Οπότε να προσθέσω ότι χθε το βράδυ, στις 10 χθε το βράδυ, ολοκληρώσαμε τον τριμερή διάλογο για τα σύρματα δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά και δικού του ανθρώπου, κύριε Επίτροπε, που ήταν ε, μαζί μα χθε το βράδυ. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό για του Ευρωπαίου πολίτε και είναι και ένα χειρό μήνυμα. Ε, το Rome like at home, δηλαδή το τηλεφωνήστε, χρησιμοποιήστε το κινητό σα όπω στην χώρα σα, χωρί τέλη ένα πολύ σημαντικό. Και θέλουμε λοιπόν διαδίκτυο υψηλή ταχύτητα, υψηλή ποιότητα, διαδίκτυο παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δωρεάν. Με δωρεάν πρόσβαση και αυτό είναι πολύ σημαντικό από την οπτική μας γωνία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά επί του θέματος. Ελπίζω και ότι το Συμβούλιο θα συμφωνήσει και αυτό για ένα καλό αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Ξεκινάει η συζήτηση. Κυρία Καστίγιο, από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε που παρασβήσχεστε για μία ακόμα φορά εδώ στην Επιτροπή μας. Τώρα, εδώ ε, βρισκόμαστε αν θέλετε στην ε, τελική πορεία αν θέλετε σε ό,τι αφορά τη θητεία μας. Οπότε ε, εκείνο που ε, είναι πραγματικότητα είναι ότι έχουν επιτευχθεί πάρα πολλά σε αυτό το τομέα ε, έτσι ώστε να έχουμε την εντύπωση ότι η όλη διαδικασία ξεκίνησε τέσσερα χρόνια πριν. Υπήρξαν δηλαδή 21 διαφορετικά νομοθετήματα και 30 συνολικά πρωτοβουλίε, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων αυτών των νομοθετημάτων για να ε, επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Με βασικό δηλαδή στόχο να προωθήσουμε την νέα ψηφιακή αγορά. Γιατί ακριβώ αυτή η νέα ψηφιακή αγορά είναι εκείνη που θα μα ε, βοηθήσει να ε, διέλθουμε αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό προκειμένου η ευρωπαϊκή κοινωνία και η οικονομία να μπορέσει να αξιοποιήσει όλες αυτές τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ψηφιακή επανάσταση. Πολλά λοιπόν έχουν ολοκληρωθεί και τώρα βρισκόμαστε σε φάση επίτευξη περαιτέρω προόδου σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τον κανονισμό για τον ένισα, τα ζητήματα ε, δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία και ούτω καθεξή. Ε, και από εκεί και μετά, βέβαια, ζητήματα συνδεσιμότητα και ούτω καθεξή. Άρα λοιπόν, τώρα δύο κύριε επιτυχέ οι οποίε είναι απαραίτητε, οι οποίε αν θέλετε θα βάλουν τις τελευταίες πινελιές εντό εισαγωγικών σε αυτό το σύστημα που έχουμε δημιουργήσει. Ποια είναι αυτά, η νέα στρατηγική για την, ε, ε κυβερνο, ε, για την κυβερνοασφάλεια, πολύ σημαντικό το ε, αναφέρατε κι εσείς, η τελευταία δηλαδή η στρατηγική είχε υιοθετηθεί το 2013, αν δεν απατώμε, και βέβαια αυτό σημαίνει ότι σε τέσσερα χρόνια πολλά έχουν αλλάξει στον κόσμο μας. Και δεύτερο στοιχείο η ελεύθερη ροή των δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, free flow of data. Είναι αυτή η ελεύθερη ε, ροή απολύτως απαραίτητη προκειμένου να δράξει τις ευκαιρίες που έχει μπροστά της Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά από στοιχεία που καταδεικνύουν ότι εάν υπάρξει κατάλληλη νομοθεσία σε ε, μια σειρά από τομείς, για παράδειγμα συνδεσιμότητα, αλλά ειδικότερα ελεύθερη ροή των δεδομένων, η ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία, ειδικότερα για παράδειγμα ο τομέας τη μεταποίηση ή για παράδειγμα αν σκεφτούμε το βιομηχανικό λογισμικό και τον ηγετικό ρόλο που καταλαμβάνει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν λοιπόν, μπορούν να αποτελέσουν ε, να δώσουν τι δυνατότητε να αποτελέσουμε παγκόσμιο ηγέτη, ο δικό μα κλάδο δηλαδή, ε, αφού και το Internet of Things, το δίκτυο δηλαδή το διαδίκτυο των πραγμάτων, έχει μεταβάλει τελείως το μοντέλο του ποιες είναι οι πηγές των δεδομένων, από πού προέρχονται. Προσωπικά δηλαδή δεδομένα, ε, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και ούτω καθεξής, αλλά τώρα έχουμε και νέα δεδομένα, από μηχάνημα σε μηχάνημα, μεταξύ δηλαδή των ε, πραγμάτων του διαδικτύου των πραγμάτων. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μοναδική ευκαιρία να καταστεί ηγέτης σε ό,τι αφορά την παγκόσμια οικονομία των δεδομένων. Άρα λοιπόν, σε σχέση με αυτό το ζήτημα θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω, θα υπάρξει πρόταση από τη δική σας ε, πλευρά ε, για αυτήν την ελεύθερη ροή των δεδομένων. Μια πρόταση την οποία πραγματικά αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, αναφέρεται κάτι το τρομακτικό, ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος της θητείας μας. Αλλά έχετε δίκιο σε δύο χρόνια θα υπάρξουν νέε εκλογέ, οπότε θα πρέπει να ολοκληρώσουμε όλε τι δραστηριότητε που έχουμε ξεκινήσει και οι οποίε σχετίζονται με την ενιαία ψηφιακή αγορά. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια πρέπει να τι ολοκληρώσουμε. Η κυρία Κουπούλα Νάτρη τώρα, εκ μέρου των Σοσιαλιστών, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ε, εκτιμώ το γεγονό ότι έχει ε, ενδιαφερθεί πάρα πολύ για αυτά τα ζητήματα ο Αντιπρόεδρο ε, και ε, καλωσορίζουμε εδώ και τον, ε, ε, τον όμιλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ελπίζουμε να έχουμε μια πολύ χρήσιμη συνεργασία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά της ψηφιακής οικονομίας. Πάντως, εδώ το ζήτημα είναι η ψηφιακή οικονομία και η κοινωνία ε, παρότι η ονομασία εδώ που χρησιμοποιούμε είναι η νέα ψηφιακή αγορά. Ίσως δηλαδή στο πλαίσιο της επόμενης επιτροπής να δοθεί μια διαφορετική ονομασία σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο την ψηφιακή αγορά. Εάν δηλαδή δεν επιτύχουμε κάτι ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο πεδίο της ψηφιοποίησης, πραγματικά δεν θα επιτύχουμε αυτά που ε, ε, επιθυμούμε και δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καινοτοπίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Αμερικανική Ήπειρο, ε, στην Ασία και ενδεχομένω κάποια στιγμή και στην Αφρική. Αυτό θα σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα μπορέσουμε ανταποκριθούμε σε οικονομικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε την υποδομή μας, θα πρέπει να ενημερώσουμε τις, δεξιότητέ τις δεξιότητες μας και από εκεί και μετά να φροντίσουμε οι καινοτομίες μας να βρίσκουν πρόσβαση στην αγορά. Μόνο τότε θα μπορούμε να κάνουμε λόγο για ενιαία ψηφιακή αγορά. Ας δώσουμε λοιπόν περισσότερη έμφαση, περισσότερη προτεραιότητα στην ε, δημιουργία και την καινοτομία. Πράγμα το οποίο βέβαια αποτελεί αρμοδιότητα του συνόλου της Επιτροπής και όχι μόνο του Αντιπροέδρου Άνσιπ, αλλά είναι σημαντικό. Δηλαδή καινοτομία. Ο ρόλος της καινοτομία για να δημιουργήσει νέα στοιχεία στην οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κοινωνία, το ψηφιακό χάσμα, digital divide που αναφέρατε, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και δηλαδή στον κώδικα τον οποίο εμείς προετοιμάζουμε τώρα, η Επιτροπή αναφέρει ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία ε, δεν ε, βρίσκονται, δηλαδή δεν έχουν προχωρήσει όσο άλλα. Ενώ άλλα κράτη-μέλη λένε ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά όλοι μα θα πρέπει να εξεχρονίσουμε τι υποδομέ μα και να μην ε, παρκούμαστε σε παροχημένε υποδομές οι οποίε υπήρχαν πριν από δεκαετίες ήδη. Όπου δηλαδή υπάρχουν κανονιστικά υποστηρικτικά μέτρα ή χρηματοδοτικά μέτρα ή οτιδήποτε άλλο, πάντοτε θα πρέπει να στοχεύουν στην αξιοποίηση των πλέον αποτελεσματικών και σύγχρονων τεχνολογιών. Επίσης ε, και ε, εσείς ε, κύριε την Πρόεδρε και οι συνάδελφοι Μιλάγιο και Καστήλιο αναφέρθηκαν στα ζητήματα της κυβερνού ασφάλειας. Προφανώς αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Αλλά πρέπει να δούμε και ποια είναι τα κονδύλια τα οποία μπορούμε να συγκεντρώσουμε για αυτόν τον σκοπό. Εδώ δηλαδή βλέπουμε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές και προσεγγίσεις ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Καλό είναι όμω ε, το γεγονό ότι δηλαδή δεν είναι όλα, δεν λαμβάνουν όλα χώρα σε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχει το κέντρο για την ε, ψηφιακή ασφάλεια στη δική μου χώρα, ε, στο οποίο συμμετέχουν διάφορα κράτη-μέλη, παρότι δεν εντάσσεται στο... στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, γιατί ε, πολλέ φορέ βλέπουμε τα κράτη-μέλη να ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε τέτοιε πρωτοβουλίε όταν δεν είναι υποχρεωτικέ, δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του, όταν δηλαδή δεν εντάσσονται στο στενό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά τώρα την ιδιοκτησία των δεδομένων, το ownership. Ε, ε, έχει κάτι έτοιμο, η Επιτροπή ετοιμάζει κάτι. Δεν έχω δηλαδή μια γνώμη ως προς το κατά πόσο θα πρέπει να ρυθμίσουμε κανονιστικά αυτό το τομέα ή όχι. Αλλά ε, σίγουρα σε μια κοινωνία η οποία βασίζεται στα δεδομένα θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση του ζητήματος της ιδιοκτησίας της κατοχής των δεδομένων. Τέλος, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της περιαγωγή του roaming ε, έγινε αναφορά από την Επιτροπή αυτό που ακούμε είναι ότι πολλές εξαιρέσεις, ε, αιτήματα εξαίρεσης αποστέλλονται στις ε, εθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι επιχειρήσει πάροχοι δηλαδή των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ε, αναφέρουν ότι δεν είναι σε θέση ακόμα να εφαρμόσουν αυτές τις αυτή την κατάργηση τη περιαγωγή. Δηλαδή, σε πολλέ περιπτώσει δεν θα είναι δυνατό να παράσχουν απόλυτα δωρεάν ε, υπηρεσίε περιαγωγή. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτέ τι περιπτώσει, σε αυτέ τι εξαιρέσει, 85% ε, ε, της ε, τιμής. Δηλαδή, από τα 50 ευρώ ανά γιγαμπίτ τώρα έχουμε φτάσει στα 7,7. 85 λοιπόν της εκατό μείωση ακόμα κι αν ή ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υπάρχει πλέον μηδενική χρέωση περιαγωγής. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, Συνάδελφα, αναφερθήκατε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και ίσως στην ακρόαση που θα κάνουμε πλευρά του Κοινοβουλίου ε, μαζί με την Επιτροπή ΚΑΛΤ ε, θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε αυτό στη νέα δηλαδή οριστήσα επίτροπο που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας που θα λάβει χώρα 20 Ιουνίου. Ναι, ημερομηνία που δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, αλλά μάλλον θα είναι το 20 Ιουνίου το απόγευμα. Είναι απολύτως απαραίτητο να παρευρεθούμε εκεί, μαζί με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Πολιτισμού. Και είναι εξίσου απαραίτητο να ε, προετοιμάσουμε λίγο τι ε, ερωτήσεις των συντονιστών από την πλευρά των ε, πολιτικών ομάδων. Τρει ερωτήσει θα τεθούν από την ΙΤΡΕ, τρει ερωτήσει θα τεθούν από την Επιτροπή Πολιτισμού και από εκεί και μετά έως 25 συμπληρωματικά ερωτήματα σε ό,τι αφορά ε, που θα τεθούν στην ορθήσα ε, επιτροπή. Ο κύριος Κρανσοντεύσκη ε, έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποιες συγκεκριμένε ερωτήσεις. προς τον κύριο Πίτροπο για το θέμα των πραγματικών δικαιωμάτων στο ψηφιακό πλαίσιο, στο πλαίσιο ψηφιακής αγοράς. Ξέρω ότι συμφωνούμε για κάποιους γενικούς όρους και κατηγορίες, αλλά με έκπληξη είδα αυτή να αφορά σε κάποια ισορροπία όσον αφορά στόχους και συμφέροντα στην ψηφιακή αγορά. Ξέρετε ποια είναι τα επίμαχα ζητήματα εδώ το text data mining και άλλα ζητήματα. Καμιά φορά όμως πρέπει να σας πω ότι έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν καθοριστεί σωστά μέχρι τώρα όλοι οι όροι και οι έννοιες σε αυτό το τομέα. Και αυτό είναι δύσκολο ας πούμε να οριστεί. Καμιά φορά Παραδείγματο χάρη έχουμε προβλήματα όπω ποια είναι η ενεργητική και ποια είναι η παθητική πλατφόρμα, ας πούμε, τα platforms. Ο Επίτροπος ξέρει, α πούμε, ακριβώς μια διαφορά μεταξύ μια ενεργούς και μιας παθητικής πλατφόρμας. Γιατί είναι δύσκολες αυτές οι έννοιε καμιά φορά. Και εσείς, Επίτροπε, προσπαθείτε να δημιουργήστε μια ακριβέστερη έννοια και ορισμό σε αυτό το θέμα ώστε να βοηθήσετε και εμάς που ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Αυτό το λέω έτσι ενδεικτικά. Έχουμε και άλλα ζητήματα παρόμοια. για τα οποία και οι ίδιοι οι νομικοί και οι εμπειρογνώμονες δεν έχουν ξεκάθαρη ιδέα για το τι σημαίνουν αυτές οι έννοιες και οι όροι. Και πάλι, ενεργός και παθητική πλατφόρμα, ας πούμε, τι, διαφορά έχει το ένα από το άλλο και πώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε καλύτερα τις έννοιες και τους όρους αυτούς. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, για τα σχόλια, λέει ο πρόεδρο. Ε, Κόκλιτσεκ, επόμενος ομιλητής, εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο απλές ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τα προγράμματα δεδομένων. Κούκκις και τα λοιπά. Εδώ πώς μπορούμε να έχουμε κάποια προστασία. Γιατί, εντάξει, μπορείτε να κάνετε προγραμματισμό, μπορείτε να προετοιμάσετε αυτά τα προγράμματα, κάποια είναι σε Excel κιόλα, αλλά κάποια άλλα μπορείτε να τα κάνετε μόνο σας. Και συνεχίζοντα την ερώτηση του αγαπητού συναδελφού προηγουμένω, ποια είναι η διαφορά μεταξύ απλού προγραμματισμού που θα πρέπει εντάξει να έχει κάποιο είδο προστασίας, αλλά και μεταξύ αυτού λοιπόν και κάποιο άλλο στοιχείο όπως ένα πολύ προχωρημένο κούκι ας πούμε, πρέπει να έχει άλλο επίπεδο προστασίας. Μετά η κάλυψη. Αν πάτε σε διάφορες χώρες, είτε είναι η Αυστρία, η Τσεχία, η Γερμανία, ακόμα και στους αυτοκινητόδρομους ή στα τρένα, θα δείτε ότι δεν υπάρχει σήμα σε πολλά μέρη. Ανεξαρτήτως χώρας, έτσι το ξαναλέω. Οπότε, εδώ μιλάμε για μια ανάγκη που αφορά όλες τις χώρες ώστε αυτές να διασφαλίσουν υψηλής ταχύτητας δεδομένα επίγεια και την διάθεσή τους όχι μόνο δηλαδή σε επικοινωνικοδικημένες περιοχές, αλλά κυρίως σε διάφορους κόμβους μεταφορών, ακόμα και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πάμε σε μία όπου το σήμα είναι πολύ αδύναμο ή μηδενικό. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτό να το καλύψουμε. Αυτά είναι τα δύο ερωτηματά μου. Uh, thank you very Ευχαριστώ, συνάδελφε. Να ρωτήσω κι εγώ. Κάτι άλλο, όχι, πρώτα κύριο κύριος Μπλάνκο Λόπε. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, γίνεται λόγο για πνευματικά δικαιώματα και τη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα ήθελα να μας πείτε αν θα προτείνετε αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των κανόνων πραγματικών δικαιωμάτων που απομακρύνονται από αυτό το στόχο. Εξάλλου μόλις ψηφίσαμε μία έκθεση μαζί με την ΙΝΚΟ για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση η Κομισιόν λέει ότι θα αναλάβει δράση σε σχέση με την ε, σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και πλατφορμών που βλέπουν και ένα νομικό εργαλείο. Θέλετε να μας πείτε ποιο θα ήταν αυτό το νομικό εργαλείο σε σχέση με την ευθύνη μεσαζόντων και πότε θα παρουσιάσετε αυτήν την πολυδιαφημισμένη, αυτό το πολυδιαφημισμένο οδηγό. Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε κάτι για τα ευρυζωνικά δίκτυα και την εφαρμογή τους. Είχαμε πει ότι θα πρέπει ετησίως να χρηματοδοτούνται 7 με 12 προγράμματα μέχρι το 22. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για περιοχές όπως η δικιά μου η Γαλλικία με μεγάλα κομμάτια υπαίθρου τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα φυγή πληθυσμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριος, η κυρία Βερκούνα λέει ο πρόεδρος. Ναι πρόεδρε ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ανσίπ γιατί νομίζω ότι ήταν πολύ ενεργητική η Κομισιόν πρόσφατα για αυτό το θέμα και όπως είπατε και εσείς, υποβάλατε πολλές ε, προτάσεις τα τελευταία χρόνια και μήνες και τώρα είναι η σειρά του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου να πάρουν αποφάσεις και να αρχίσουν εφαρμογή αυτών των αποφάσεων οι χώρες μέλη. Ξέρετε όλοι ότι αυτό είναι ένα κλειδί για την επιτυχία μας στο μέλλον, ότι θα πρέπει δηλαδή να είμαστε ανταγωνιστικοί στον ψηφιακό κόσμο επίσης. Πείτε μου λοιπόν Ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη αν προσεγγίσουμε το ψηφιακό κόσμο παγκοσμίω, Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία, θεωρείτε ότι είμαστε αρκετά γρήγοροι και ανταγωνιστικοί ή είμαστε κάπως αργοί. Έχουμε πολλή γραφειοκρατία και αργή διοίκηση σε σχέση με τον ψηφιακό κόσμο. Επίσης, αν θα έπρεπε να επιλέξετε δύο-τρία πεδία για να είμαστε πιο ενεργοί στον ψηφιακό κόσμο στην Ευρώπη, αυτά ποια θα ήταν και ποια θα ήταν σημαντικά βήματα που θα έπρεπε να κάνουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ο κύριος Κολομπάτσεφ λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Μπουζέκ. έχουμε μια πρόταση από τη χώρα μου για τις 20 του Ιούνιου. Η ερώτησή μου προς τον κύριο Άνσιπ αφορά τον κανονισμό για την ιδιωτική ζωή, το e-privacy. Όπως ξέρετε, έχουμε το GDPR και θα ισχύσει από τις 25 Μαΐου του 2018. Η πρόταση όμω για την ηλεκτρονική ιδιωτική ζωή τη Κομισιόν, το e-Privacy, αφορά την ίδια ημερομηνία. Για το GDPR, βέβαια εντάξει, θα έχουμε ξεχωριστή νομοθεσία, οπότε μπορεί να υιοθετηθεί νωρίτερα. Αλλά γιατί την ίδια μέρα. Αν κάνουμε μια αναβολή, εντάξει, να μην το αναβάλουμε για πολύ κατηραλιστικό. έξι μήνες ε, ας πούμε. Αλλά μην πάμε πέρα του ορίζοντα των εργασιών του Κοινοβουλίου ή τη Κομισιόν. Ξέρετε ότι έχουμε και άλλα επίμαχα, μάλλον πολλά επίμαχα ζητήματα στον τομέα τη ηλεκτρονική ιδιωτικής ζωή. Ήδη μίλησε ένα αδόφο για τα cookies, ας πούμε, για browsers, για gatekeepers, κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, τις ε, ε, της εταιρείε τηλεπικοινωνιών σε σχέση με κάποια λογισμικά. Ήδη έχουμε λοιπόν πολλά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε Ευτυχώς τουλάχιστον έχουμε έναν έμπειρο εισηγητή, η κυρία Λαουριστίν. Αν όμως έχουμε χρόνο για συζητήσεις, να προσπαθήσουμε να μην το αναβάλουμε για πολύ, τρεις με έξι μήνες το πολύ καταρχάς και κατά δεύτερον, να δώσουμε αρκετό χρόνο στις επιχειρήσεις, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις της νέας πρωτοβουλίας και του νέου κανονισμού που ενδεχομένως θα πρέπει να προβλέπει νέο λογισμικό αν ας πούμε κάνετε browsers ε, δεν θα πρέπει να καθίσετε πάνω από τρει μήνες. 25 Μαΐου όλα θα πρέπει να εφαρμοστούν αργότερα, 25 Αυγούστου, τρει μήνες, όχι παραπάνω λοιπόν. Θα πρέπει λοιπόν ο κανονισμός να παρέχει επαρκή χρόνο και μετά θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να γίνεται με το λογισμικό σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού, το πολύ να έχουμε μια αναβολή δηλαδή 6 με 9 μήνες. Αυτά σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, με το χρονισμό, το timing για την ιδιωτική ηλεκτρονική ζωή. Ευχαριστώ συνάδελφε ο και εγώ να προσθέσω μια ερώτηση γενική φύση στον Αντιπρόεδρο. 70 80% της καινοτομίας στην οικονομία πετυχαίνεται στον ψηφιακό τομέα ή προέρχεται εδώ πάντων να βάλει χώρα στο ψηφιακό τομέα. Υγεία, ας πούμε στις εχειρήσει χάρη στα συστήματα τα οποία είναι σωματωμένα, υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια και έχουμε θαυμάσια αποτελέσματα. Το ίδιο ας πούμε στην αγορά ενέργειας. το ευφυές ε, δίκτυο, οι ευφυείς ε, μετρητές. Όλα αυτά γίνονται χάρη στα ψηφιακά συστήματα. Και μεγάλο ρόλο εδώ στην καινοτομία παίζουν και οι startups. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να χρηματοδοτήσουμε και να επενδύσουμε στις startups. Γιατί οι επενδυτές ενδιαφέρονται για αυτές τις επιχειρήσεις στην Αμερικανική αγορά και όχι στην Ευρωπαϊκή. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για τις αγορές στο Μιλάνο, Βερολίνο, στο Λονδίνο, Βαρκελόνη. Για επιχειρήσεις που έχουν στόχο την παρουσία στην Αμερικανική αγορά και την ε, προσέλκυση επενδύσεων από εκεί. Εντάξει, ξέρω ότι είναι κάπως περίπλοκο ή δύσκολο αυτό το θέμα, αλλά θα αρχίσουμε να το εξετάζουμε. Θέλουμε να είμαστε καινοτόμοι για το μέλλον και θέλουμε να πετύχουμε πρόοδο στην ενιαία ψηφιακή αγορά και μέσω της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ένωσης θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ενισχύσουμε τις startups. Γενική φύση ερώτηση αυτή, έτσι, αλλά στο σκεφτούμε. Τώρα για τα υπόλοιπα, κύριε Αντιπρόεδρε, παρακαλώ έχετε το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, για τις ερωτήσεις, για τις προτάσεις. Επιτρέψτε μου όμως καταρχάς ένα γενικό σχόλιο. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που η Βουλγαρία όρισε την νέα επίτροπο. Ξέρετε, είχα πολλούς φακέλους, πολλά θέματα στα χέρια μου. Και ελπίζω ότι η Μαρία θα πετύχει στην ε, ακροασή τη ε, ενώπιον και της δικής σας επιτροπής, η νέα η πρωταθήσα επίτροπος από τη Βουλγαρία. Εγώ είμαι βέβαιος ότι είναι πολύ καλή η Επίτροπος Ψηφιακής Αγοράς. Να ευχαριστήσω με την ευκαιρία κυρία Τικαστήγιο για όσα κάνατε για την ενιαία ψηφιακή αγορά πήγαμε μπροστά σε αυτόν τον τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ήδη είμαστε κοντά σε, μια, σε αυτό που ονομάζουμε ενιαία ψηφιακή αγορά. Ε, ως προς τα τέλη περιεγωγής, όπως είπα, η ημερομηνία κλείνει είναι 15 Ιουνίου. Πάντως, δεν ε, έχουν καταφέρει όλοι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας να παράσχουν αυτή την υπηρεσία, τη δωρεάν περιοχή. Το να τηλεφωνείς δηλαδή όπως όταν είσαι στη χώρα σου για τις ε, εταιρείε, για τους παρόχους που θα έχουν δυσκολίες. Ξέρουμε, για παράδειγμα, στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν γενναιόδωρα πακέτα και σχετικά φθηνές υπηρεσίες. Εκεί μπορεί να χρειάζεται να υπάρξει ένα όριο στην δωρεάν περιοχή, και αυτό δεν αποτελεί, μπορεί να αποτελεί πρόσχημα να αυξηθούν οι τιμές για τους χρήστες οι οποίοι δεν πρόκειται να ταξιδέψουν ποτέ σε κάποια άλλη χώρα. Ο Πιλάρ Καστίγιο όμως ανέφερε και το θέμα της ασφαλείας των κυβερνοχώρων, της ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για μένα το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ πολύ σημαντικό το είπα και στην εισαγωγή μου. Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε να θέσουμε προδιαγραφές ασφαλεία για το διαδίκτυο των πραγμάτων, για τα botnets και άλλο κακόβουλο λογισμικό το οποίο ε, επιτίθεται κατά μεγάλων επιχειρήσεων, παρόχων υπηρεσιών κλπ. Στις ΗΠΑ, ξέρετε, το ίντερνετ των πραγμάτων, όπως το λέμε, είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και γενικότερη ασφάλεια των ηλεκτρονικών επιχειρονιών. Όσοι κατασκευάζουν, ας πούμε, λάμπες, για παράδειγμα, φθηνές συσκευές, συσκευές που είναι φθηνές γενικά, αλλά είναι συνδεμένες με το διαδικτύο, αυτοί δεν προσέχουν και πολύ τα θέματα της ασφάλειας, της κυβέρνων ασφάλειας. Όμως στους χώρους όπου ε, διακυβεύεται η κυβερνοσφάλεια και εκεί βλέπουμε ότι πολλοί κόσμοι δεν νοιάζεται. Ας πούμε, δείτε τι γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα, με τις ταμπλέτες. Ε, κάποιοι επαγρυπνούν, αλλά οι περισσότεροι όχι. Φυσικά θα αλλάξουν αυτά. Θα πρέπει όλοι να αλλάξουν τις βασικές τους ρυθμίσεις. Αλλά έχουμε και συσκευές όπως πάρτε μια ηλεκτρική σκούπα για παράδειγμα. για οικιακή χρήση. Ποιος θα κάτσει να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις αυτής της συσκευής. Γι' αυτό και οι κακοί εντό εισαγωγικών δημιουργούν Bottlenecks. Αξιοποιώντας ακριβώς τις διασυνδεμένες συσκευές. Τις συσκευές που επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε να προκρίνουμε προδιαγραφές ασφαλείας αλλά και γενικότερα να παγρυπνούμε, να είμαστε πιο προσεκτική ε, στην, την την υγιεινή του διαδικτύου. Γιατί όλοι πλένουμε τα χέρια μας για λόγους υγιεινής, ναι, αυτό το ξέρουμε, το έχουμε συνηθίσει, το κάνουμε. Είναι πολύ πιο δύσκολο όμως όταν το πράγμα αφορά διασυνδεδεμένε συσκευέ μέσω διαδικτύου. Εκεί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα σκεφτόμαστε. Το διαδίκτυο των πραγμάτων, όπως τη λέμε, ε, θα φορά σε λίγο καιρό συσκευές όπως είπα μια ηλεκτρική σκούπα, ένα ψυγείο, αυτές οι συσκευές. Ένα σίδερο για παράδειγμα. Όταν ας πούμε κάποια συσκευή τραβάει πολύ ρεύμα μπορεί το ψυγείο να λειτουργεί σε υψηλότερη θερμοκρασία για να αποφύγουμε τι εχμές κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό γίνεται μέσω διαδικτύου με τι ευφυείς συσκευέ. Όταν εγώ σιδερώνω μπορεί το ψυγείο να μην ψύχει τόσο πολύ, να μην χρειάζεται να ψύχει τόσο πολύ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ίσω και 100 εκατομμύριων το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει λοιπόν ένα νόημα να συνδέει κανεί να διασυνδέει κανείς το ψυγείο με το σίδερο, αλλά αυτό έχει και κινδύνους. Εκεί λοιπόν θα χρειαστεί να τροποποιήσουμε κάποιες ρυθμίσεις για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Θα το έλεγα είναι κυβερνό υγιεινή αν θέλετε, αν με επιτρέπει το όρος. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια γενικότερη στρατηγική και αν πρόκειται για στρατηγική πρέπει και η ΕΝΗΣΑ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Προστασία και την Ασφάλεια των Δεδομένων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών να Δηλαδή μια νέα εντολή. Ο λοιπόν πρέπει να ενεργοποιηθεί. Αποτελεί ένα κέντρο αριστείας, το οποίο γίνεται όλο και καλύτερο. Χρειαζόμαστε όμως, όμως και άλλα τέτοια κέντρα αριστείας για την κυβερνοασφάλεια. Πρέπει να αντεπεξέλθουμε στις ε, απειλές όπως κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα η θέση μας είναι εν μέρη επισφαλής. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα για την ασφάλεια, αλλά όχι όσα θα έπρεπε. Τώρα για τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες, όπως προείπα. Κάποιες μεγαλύτερες χώρες δεν ασχολούνται πολύ με το θέμα με τη συνεργασία δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί τα καταφέρνουν μόνες τους. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο η είναι <laughs> τα μικρότερα κρατημέλη να αποτείνονται για συνεργασία για την βελτίωση επιχειρησιακών δυνατοτήτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώ. να, άλλο ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Έτσι όπως το βλέπω το πράγμα, χρειαζόμαστε επιχειρησιακές δυνατότητες για να αντιμετωπίσουμε τις κυβερνοαπειλέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, ελεύθερη ροή, ανταλλαγές στοιχείων, δεδομένων. Άλλο ένα ωραίο θέμα. Πέρσι τον Δεκέμβριο, στο Συμβουλίο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών, ζήτησε με το θέμα. 20 έλαβαν τον λόγο. Οι 18 ζήτησαν άμεση δράση, άμεση κινητοποίηση και σε νομικό επίπεδο και σε νομοθετικό αν θέλετε επίπεδο. Ένας είπε γιατί όχι, ναι, ένας είχε τις εμβολίες του αλλά φαίνεται ότι όλοι θα υποστηρίξουν την αρχή της ελεύθερης ανταλλαγής δεδομένων. Όπως είπα, ένας μόνο υπουργό ήταν κατά. Επεκτείναμε την θέση μας για να καλύψει, να συμπεριλάβει αν θέλετε και εγγυήσεις στο πλαίσιο της πρόσβασης στοιχείων, δεδομένων που είναι σε κάποια άλλη χώρα. Θεωρώ ότι με την παροχή εγγύσεων και ο τελευταίος υπουργός που είχε ε, θα συμφωνήσει μαζί μας. Γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ισχύουν 56 διαφορετικές νομοθεσίες ή σύνολα κανόνων σε 21 χώρες και αυτή είναι η τάση ξέρετε παντού σε ολόκληρο τον, τον κόσμο οι μεγάλες χώρες το ξαναλέω αντιπεξέρχονται σε μια κατακριβατισμένη Ευρώπη γιατί μπορούν να έχουν την πολυτέλεια να διαθέτουν 28 κέντρα δεδομένων σε 28 χώρες. Αλλά τι γίνεται με τις μικρομεσαίες, τι γίνεται με τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν μπορέσουν ποτέ να δημιουργήσουν 28 κέντρα δεδομένων σε 28 κράτη-μέλη. Άρα ποιο είναι το μήνυμα, τι βγαίνει από όλα αυτά. Τι θα πούμε στους ανθρώπους μας. Θα πούμε πηγαίνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε μια κατακρεματισμένη αγορά. Η Αμερική στέλνει το μήνυμα. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πω στου ανθρώπου μα, στου πολίτε μα, μην σπίτι μην κάνετε τίποτα. Όχι, ξεκινήστε, βγείτε και επιχειρήστε. Τον Σεπτέμβριο ελπίζω ότι στο θέμα της ελεύθερη ανταλλαγή στοιχείων θα έχουμε μια έτοιμη νομοθετική πρόταση και ότι μετά από λίγο θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με τα θέματα της διοκτησία των στοιχείων, των δεδομένων, τα θέματα της πρόσβασης, τα θέματα της ε, νομικής ευθύνης. Για να είμαι ειλικρινής, η Κομισιόν δεν είναι έτοιμη. Δεν έχουμε ε, κατεβάσει πρόταση για το θέμα της διοκτησίας των δεδομένων. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο. Ε, κατά τα άλλα, συμφωνώ με όσους υποστήριξαν ότι η αρχή αυτή είναι πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Είχαμε συμβούλιο ανταγωνιστικότητας προχθές. Ε, κανείς δεν ε, είχε αντίρρηση με την ανταλλαγή δεδομένων. Οι περισσότεροι υποστήριξαν και πάλι την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, για την ιδιοκτησία και πάλι των δεδομένων. Ποιε είναι οι σχετικέ πρακτικέ. Ξέρετε, οι πρακτικέ διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για κάποιε επιχειρήσει η ιδιοκτησία των δεδομένων δεν είναι σημαντική. Καθόλου σημαντική. Θέλω απλώ πρόσβαση στα δεδομένα. Για παράδειγμα, η Σκάνια συνέδεσε, διασυνέδεσε 230.000 φορτηγά σε όλη την Ευρώπη. Ε, είπαν, εμάς δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ιδιοκτησία αυτών των δεδομένων. Εμείς, λένε, θέλουμε απλώς να τα αξιοποιούμε. Οι Siemens το ίδιο θέλουν να αξιοποιούν τα δεδομένα, να έχουν ε, χρήση των δεδομένων. Μια άλλη όμως επιχείρηση λέει, εγώ τα θέλω δικά μου. Δεν λέω τι είναι καλύτερο και τι είναι χειρότερο. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αξιοποίηση των δεδομένων. Και εν τέλει πρέπει να εναρμονίσουμε αυτές τις προσεγγίσεις, τις μεθόδους. Κάπου πρέπει να καταλήξουμε, αν πάση περιπτώσει. Για τα θέματα της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είστε ενδεχομένω η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, αλλά σύμφωνα με αυτού που είπαν ότι είναι ε, δύσκολο να εξασφαλίσουμε έναν λογικό συγκερασμό μεταξύ των δισταμένων συμφερόντων. Εμείς με την πρότασή μας θέλουμε να εξασφαλίσουμε ισορροπία να συνδυάσουμε δίσταμενα συμφέροντα αλλά πάντα κάποιος θα είναι δυσαρεστημένος ξέρετε τώρα με την πρότασή μας για τα πνευματικά διανοητικά δικαιώματα θέλουμε την αρχή της χώρας προέλευσης να την επεκτείνουμε και να θεσπίσουμε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων. Ο στόχος μας είναι με άλλα λόγια να διπλασιάσουμε τον όγκο του περιεχομένου, ο οποίος ήταν προσβάσιμος πέραν των συνόρων, διασυνοριακά για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σήμερα το διοικητικό κόστος για τη χωρίση άδεια χρήση αυτών των δεδομένων είναι πολύ ψηλό. Πολύ ψηλό, πάρα πολύ ψηλό. Και αυτό αποτελεί και εμπόδιο για τον απλό Ευρωπαίο πολίτη που θέλει να δει μια ταινία όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό. Οι πάροχοι δεν θέλουν να αναλάβουν το κόστος αυτό και αυτό είναι πρόβλημα και για τους δημιουργούς. Δηλαδή δεν θα αμείβονται ικανοποιητικά εάν το θέμα της ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων παραμείνει ασαφές. Αν δηλαδή λόγω των γνωστών εμποδίων ο κόσμος ε, υθετεί το γκρίζες μεθόδους, παράνομες μεθόδους για να αποκτήσει πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο. Όπως γνωρίζουμε, σύμφωνα με μετρήσεις, 68% των χρηστών λένε ότι έχουν κατεβάσει παράνομα περιεχόμενο. Πρόβλημα για τους ε, δημιουργούς, ίσως όχι πρόβλημα <laughs> για τους χρήστες που κατεβάζουν δωρεάν περιεχόμενο, αλλά επαναλαμβάνω, οι δημιουργοί τελικώς είναι χαμένοι. Άρα, θέλουμε καλύτερη πρόσβαση, διεθνή, διασυνοριακή πρόσβαση προς ψηφιακό περιεχόμενο. Και όταν λέω ελεύθερη πρόσβαση δεν εννοώ δωρεάν, αλλά να υπάρχει δυνατότητα, νόμιμη δυνατότητα πρόσβασης. Προτείνει μια μορφή λοιπόν ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεν λέω ότι το ενδιαφέρον είναι αντίστοιχο με, το, με τον όγκο των ανθρώπων που πηγαίνουν στο κινηματογράφο για να δουν μια ταινία, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον. Κάποιοι θέλουν να κατεβάσουν βιβλία ή ταινίε, όπω είπα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ε, στη διάθεσή του μια νόμιμη λύση. Το ίδιο για του εκπαιδευτικού σκοπού. Ένα δάσκαλο, ένα καθηγητή, ο οποίο διδάσκει και σε κάποια γειτονική χώρα. Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν θέματα δικαιωμάτων γιατί αξιοποιούν υλικό σε μια παρουσίαση που καλύπτεται από κάποια συμφωνία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Και ξέρετε τώρα, αν ένα καθηγητή ε, κατεβάσει παράνομα περιεχόμενο, μπορεί να γίνει και σκάνδαλο. Θέλουμε να διευκολύνουμε λοιπόν και δασκάλου και καθηγητές, αν και δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος για τον οποίο έχουμε δρομολογήσει την πρωτοβουλία μας αυτή, γιατί εκεί υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις. Ύστερα η εξαγωγή μεγάλων όγκων δεδομένων, data extraction, και εκεί υπάρχουν κανόνες, ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προχωρήσει. Εκεί υπάρχουν σαφείς κανόνες ε, το καθεστώς είναι πολύ φιλελεύθερο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, γι' αυτό και με έκπληξη είδα την συγκεκριτή να προτείνει ακόμη πιο φιλελεύθερους κανόνες προκειμένου. Φοβούμαι ότι έτσι θα καταστρέψουμε τα εφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία όμως αποδίδουν ικανοποιητικά, λειτουργούν ικανοποιητικά σήμερα. Θα έλεγα εδώ να επιδείξουμε μεγαλύτερη σύνεση και προσοχή. Δεν υπάρχει λόγος να καταστρέψουμε ένα καλό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο διαχειριστεί ικανοποιητικά και τα πνευματικά δικαιώματα. ηλεκτρονικά καταστήματα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες λειτουργούν με βάση συνδρομή. Οι συνδρομητές αυτοί καταβάλουν μέσω των συνδρομών τους, τους δημιουργούς, 2 ε, δισεκατομμύρια το χρόνο. Υπάρχουν όμως και πλατφόρμες, άλλες πλατφόρμες, που χρηματοδοτούνται μέσω διαφημίσεων. Αυτές οι πλατφόρμες δεν έχουν μερικές χιλιάδες μόνο συνδρομητών, έχουν εκατομμύρια αν όχι δισεκατομμύρια συνδρομητέ και τι πληρώνουν στου ε, δημιουργού. Έχουμε ένα νούμερο που λέει 643 εκατομμύρια στους δημιουργούς. Δείτε τα νούμερα, Συγκρίνεται τις δωρεάν πλατφόρμες με, με τις άλλες. Και φυσικά η δημιουργία, η μουσική είναι δυσαρεστημένη. Κάποιος ουσιαστικά αξιοποιεί περιεχόμενο για να βγάζει πολύ περισσότερα δίνοντας ψίχουλα στους δημιουργούς. Και εκεί χρειαζόμαστε μια λύση για το πρόβλημα. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάνε αυτές οι διαπραγματεύσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς, επαναλαμβάνω, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες μας να έχουν νόμιμη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα. Αυτό θέλουμε, να πετύχουμε. Και θέλουμε να αμείβονται δίκαια οι δημιουργοί. Δεν λέω ποιος στόχος είναι πιο σημαντικός και οι δύο στόχοι είναι σημαντικοί. Θέλω ξαναπώ και οι δύο στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί για μένα. Τώρα, τα ε, συγγραφικά δικαιώματα ε, και τα συνεφή ε, δικαιώματα εκδοτικά είναι ένας σημαντικός τομέας και είχα ταχθεί ε, κατηγορηματικά με το μέρος εκείνων που είχαν ζητήσει μια λύση σε αυτό το τομέα. Αλλά όταν οι διάφορες δισκογραφικές εταιρείε, για παράδειγμα, είπαν ότι Ε, είχαν ε, αγοράσει για παράδειγμα τα, ε, σχετικά δικαιώματα, δηλαδή σε τους σχετικούς τίτλους, ουσιαστικά διαπιστώσαμε ότι δεν ισχύει το, το ίδιο για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις, τις εκδόσεις. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα κοινό αν θέλετε, σύστημα για όλους. Ε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά από τη μία πλευρά τον, ε, αυτόν τον τομέα, του από την άλλη εκείνο τον, ε, το δημοσιογραφικό, τον εκδοτικό και ό,τι καθεξής. Βέβαια, ε, από αυτόν τον κλάδο συχνά μας λένε ότι οι, αυτοί δηλαδή που δραστηριοποιούνται στον εκδοτικό τομέα, στον τύπο, εμ, δρούν περισσότερο ως πλατφόρμες διαμεσολάβησης. Ε, πάντως παραμένει δηλαδή εκρεμές αυτό το ζήτημα ε, των, των σχετικών δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση παρέρχεται γρήγορα ο χρόνος όταν τελικότερε απαντήσει. Πάντω, σε ό,τι αφορά το ερώτημα που τέθηκε σχέση με τι πλατφόρμε, είπα ευθύ εξ αρχή ότι δεν θα ακολουθήσουμε μια οριζόντια προσέγγιση ω Επιτροπή ω προ το ζήτημα των πλατφορμών. Γιατί είναι εύκολο κανεί να καταπνίξει ουσιαστικά την καινοτομία με υπερβολικά ρυθμισμένε, υπερ ε, ελεγχόμενες πλατφόρμες. Άρα λοιπόν εδώ προσπαθούμε να ακολουθήσουμε μία εξατομικευμένη περίπτωση. Ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, την αρχή notice and action, ναι, θα πρέπει να ε, παρέμβουμε εδώ ή συνεργατική οικονομία, collaborative economy και εδώ θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές μας. σε ό,τι αφορά στους αυτοκινητοδρόμους, ναι. Και εμένα δεν μου αρέσει η κατάσταση στη Λαπωνία, είτε δηλαδή βρισκόμαστε στο σουηδικό κομμάτι στο φιλανδικό κομμάτι, Υπάρχει πάρα πολύ καλό σήμα 4G. Εξαιρετικό. Αλλά ταυτόχρονα η πληθυσμιακή πυκνότητα είναι χαμηλότερη από ένα άτομο ένα ε, τετραγωνικό χιλιόμετρο. Οπότε ε, εκεί βλέπουμε εξαιρετική κάλυψη, ενώ για παράδειγμα το ξέρετε καλά όταν μεταβαίνουμε από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο ε, υπάρχουν ζώνες δεκάδων χιλιόμετρων όπου δεν έχουμε κανένα σήμα. Και δεν λέω σήμα ίντερνετ, δεν έχουμε καν τηλεφωνικό σήμα. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, στη Λαπωνία, ε, όπου δεν υπάρχει κανεί, όπου για να περάσει ένα αυτοκίνητο από το δρόμο πρέπει να περιμένει κανεί ώρε, έχουμε εξαιρετικό σήμα 4G, ενώ εδώ τέσσερι λωρίδε κυκλοφορία όλε ε, ε, γεμάτε, δηλαδή πλήρε κυκλοφοριακό χάο, χωρί να έχουμε σήμα. Ούτε καν τηλεφώνου. Άρα θα πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα και ειδικότερα όταν θα έχουμε αυτά τα αυτοοδηγούμενα, τα self-driving cars, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντολισμό και για το θέμα του σήματο. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις startups της νοφής, ε, είπα ότι το κύριο πρόβλημα είναι ο καταγερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς. Με τη δημιουργία της ενιαία ψηφιακή αγοράς υποστηρίζουμε ακριβώς και τις νέες μας αυτές τις startup επιχειρήσει, Γιατί δεν θα βρίσκονται αντιμέτωπε με αυτό το κατακαιρματισμένο με αυτή την κατακαιρματισμένη αγορά. δηλαδή το να δραστηριοποιηθούν τέτοιε νεοφυεί επιχειρήσει στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ δυσκολότερο από ό,τι για παράδειγμα στι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε θέλουμε να του δώσουμε περισσότερε δυνατότητε και θέλουμε να του υποστηρίξουμε στη δημιουργία hubs, ε, κέντρων δηλαδή επιχειρηματικών μεταξύ του και δικτύων μεταξύ των επιχειρήσεων startups. Και από εκεί και μετά βέβαια ε, την κατάλληλη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για αυτήν την ε, πολύ ευρεία και περιεκτική συζήτηση που έγινε για όλα ε, τα ζητήματα εδώ και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να σας ε, ξαναδούμε εδώ. τέθηκε ένα ερώτημα εδώ από δύο μέλη. Ε, εντάξει, απλά θα σας ε, πω να σε περιοριστούμε. Ε, έχουμε ίσως ε, καταρρύψει κάθε ρικόρ εδώ, 26 δηλαδή λεπτά σε ε, Επιτροπή για τις απαντήσεις. Εντάξει, Πρόεδρε, μου είπατε ότι δεν υπήρχε περιορισμό χρόνου. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα του e-privacy, τη ηλεκτρονική ιδιωτικότητα και τη σχέση δηλαδή με το Γενικό Κανονισμό Προστασία των Δεδομένων, σχετίζεται και με τι διαπραγματεύσει που γίνονται εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο και του Τριμερού διαλόγου και ακριβώς με βάση όλες αυτές τις συζητήσει θα φτάσουμε και κάποια στιγμή στην ε, ημερομηνία θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού. Πάντως, ανέκαθεν η δική μας ε, πρόθεση ήταν να αποφευθούν οι διαφορετικές ερμηνείες του λόγου κανονισμού στα διαφορετικά κράτη-μέλη. Ακριβώς λοιπόν ε, πρόθεσή μας ήταν να έχουμε θέση σε ε, εφαρμογή την ίδια ημερομηνία σε όλα τα κράτη-μέλη. Πάντω, για μένα, ε, κανονιστικό πλαίσιο για τα δεδομένα πραγματικά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχει δηλαδή μια οδηγία σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα, ε, αλλά η, ε, το πώ αυτή τελικά μεταφέρει και στην εθνική νομοθεσία ήταν πολύ διαφορετικό στα διαφορά 28 κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν, ε, το απόρριτο για παράδειγμα της, ε, της επικοινωνίας ε, στο πλαίσιο της, των επικοινωνιών είναι εγγυημένο αλλά όχι στο πλαίσιο των αιτητής. Οπότε εδώ τώρα προσπαθούμε με τον κανονισμό να δημιουργήσουμε ίσους όρους για όλες τις περιπτώσεις. Λέμε λοιπόν στον κανονισμό ότι το απόρριτο της επικοινωνίας θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ακόμα ε, και όταν αξιοποιείται άλλο μέσο επικοινωνίας, το οποίο δηλαδή ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί, ένα μελλοντικό μέσο επικοινωνίας. Και εκεί θα είναι προστατευμένο το απόρριτο των επικοινωνιών, η εμπιστευτικότητά τους. Και εδώ βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους παροχή των σχετικών υπηρεσιών και των Δηλαδή, ε, καλούνται οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις σχετικές, ε, τις, ποιότητα των, ε, ε, των, των σχετικών υπηρεσιών τους και δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταπολούν να διαβιβάσουν τα σχετικά δεδομένα. Και τώρα η νέα αρχή που ουσιαστικά επιβάλλουμε είναι η συνένεση του χρήστη, δηλαδή η συνένεση του ατόμου στο οποίο αφορούν τα δεδομένα για κάθε περαιτέρω χρήση, για την πώληση διαφημίσεων και ούτω καθεξής. Γνωρίζω πάντως ότι ε, η ε, δοτικοί του τύπου ε, ανησυχούν λίγο, αλλά από την άλλη πλευρά τι θα κάνουμε. Ε, τι θα γίνει με τα κούκκις για παράδειγμα. Ε, δηλαδή το 90% των ερωτηθέτων σε έρευνα που κάναμε δεν θέλουν κάθε φορά να κάνουν κλικ σε αυτά τα κουτάκια επιβεβαίωση του αν θέλουν δηλαδή να ε, ε, λαμβάνουν κούκκις ή όχι. Και σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις, σε ό,τι αφορά την ε, προστασία, δηλαδή της ε, ιδιωτικότητα, τα privacy settings, για παράδειγμα στα προγράμματα browser, περιήγησης δηλαδή του διαδικτύου, προσπαθούμε να έχουμε κατά νου δηλαδή να υπάρχει μια προεπιλογή υψηλής ασφάλειας, από εκεί και μετά να έχουν τη δυνατότητα οι χρήστες να αλλάζουν τις ενογορυθμίσεις αργότερα. Οπότε, εάν έχουμε διάφορους φορείς εδώ από τον ιδιωτικό τομέα του τύπου και γενικά, ε, οποιοδήποτε άλλος έχει να προτείνει κάτι το οποίο μπορεί να βελτιώσει τη σχετική πρόταση τη Επιτροπής, είμαστε ανοιχτοί να, να, να τα ακούσουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σα ευχαριστώ για την ε, πολύ επικοδομητική συνεργασία που έχουμε με την Επιτροπή σα. Πρόεδρος, ε, σας ζητώ πραγματικά συγγνώμη που σας πίεσα λίγο τώρα στο τέλος της ε, παρέμβασής σας. Ίσως ήταν δικό μου λάθος. Πραγματικά ήταν εξαιρετική η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ σημαντική λοιπόν η συζήτηση που έγινε σήμερα για ε, τα μέλη τη Επιτροπή μα, γιατί απαντήσατε σε μεγάλο βάθο στα ερωτήματα που σα θέσαμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. 29 και 22 Ιουνίου είναι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, ε, συνάδελφοι. Να είστε έτοιμοι και εκεί θα γίνουν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Επαναλαμβάνω, 21 και 22 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Hearing... Η ακρόαση στη μία και μισή. Σήμερα, έτσι. Την ώρα του μεσημεριανού, εξαιρετική ώρα. Για να δυνατήσετε όλοι, αφού δεν θα φάτε μεσημεριανό, για να είστε στην ακρόαση στη μία και μισή.